Uh, Καλησπέρα συνάδελφοι. Πριν περάσουμε στις ψηφοφορίες, έχω μια ανακοίνωση. Οι αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου μας γνωστοποίησαν την εκλογή του κ. Ντάνιελ Ντόρτον για να αντικαταστήσει τον κ. Φίλιπ Μπράντμπορν από τις 8 Ιανουαρίου και μετά. Και σύμφωνα με τα ισχύοντα, Ο κανονισμός προβλέπει ότι από τις 8 Ιανουαρίου και μετά εκλέγεται και επίσημα ο συνάδελφος. Τον καλωσορίζω και του τονίζω ότι μέχρι να ε, δοθεί η έγκριση των διαπιστευτηρίων του θα μπορεί να απολαμβάνει όλων των δικαιωμάτων του εφόσον έχει υπογράψει την προβλεπόμενη δήλωση συμφερόντων. Και τώρα περνάμε στις ψηφοφορίες. Πρώτη έκθεση είναι του κυρίου Φερέιρα. Ο εισηγητής έχει το λόγο για δύο λεπτά.